όπως αυτό που έχει προτείνει ο συνάδελφός μας Δάβιδ Μάρτιν. Και επίσης, χωρίς να καθυστερήσουμε, θα πρέπει να εγκρίνουμε και τις τρεις αυτές συμφωνίες. Ευχαριστούμε και τώρα από το ΕΛΚ ο κύριος Φιέλνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Επίτροπε, επιτέλους, έχουμε αυτή τη συμφωνία με την Σιγκαπούρη. Ε, θα πρέπει να ήταν απλά τα πράγματα, όμως χρειάστηκε μια δεκαετία. Και δεν έφταιγαν οι Σιγκαπουριανοί, Εμεί στέγαμε. Ε, πολλοί ήταν οι συναδελφοί εδώ στο σώμα που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να την ε, παρακολύσουν, ιδίω ό,τι αφορά τι επενδύσει, τη Συμφωνία για τι Επενδύσει και συνεχίζουν να παρακολύουν. Αυτό έχει βλάψει, έχει θίξει την ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική. Και η Σιγκαπούρη ε, δεν ε, έτυχε δίκαιε μεταχείριση. Εδώ λοιπόν πρέπει να πω ότι τη Συμφωνία αυτή τη θεωρώ καλή. Τη θεωρώ μια πολύ δυναμική οικονομία τη Ανατολική Ασία στη Σιγκαπούρη. Και νομίζω ότι αύριο θα πρέπει να τη θα πρέπει να υποστηρίξουμε την έγκριση των συμφοριών αυτών. Ε, υπάρχουν πολλοί εδώ που είναι κατά ε, από όλες τις πολιτικές παρατάξεις προσπαθούν να παρακολύσουν την πρόοδο της εμπορικής μας πολιτικής ε, με πρόσχημα την Κίνα. Είναι το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Θα πρέπει να ε, εξασφαλίσουμε ευρεία στήριξη και να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη μας στην όλη διαδικασία. Ευχαριστούμε και τώρα η κυρία Νίνα Γκίλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε Επίτροπε. Είμαι μέλος της αντιπροσωπείας με τις, των σχέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση χωρών ΑΖΕΑΝ. Και θεωρώ ότι οι χώρε αυτέ μπορούν να προσφέρουν πολλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχα την ευκαιρία να, συζητήσω, να συζητήσω τη συμφωνία αυτή με μια σειρά από ε, συνομιλητέ τη Σιγκαπούρη, με κυβερνητικέ οργανώσει, εκπροσώπου ανεξάρτητων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Όλοι θέλουν μια ισχυρότερη σχέση συνεργασία, εταιρική σχέση μεταξύ ε, ημών και ημών. Θεωρούμε ότι το διεθνέ εμπόριο βρίσκεται σε κατάσταση μεταβαλλόμενη οι Ηνωμένε Πολιτείε ξαναγράφουν ε, παλιού κανόνε που ήταν παγιωμένοι. Δεν είναι αξιόπιστο εμπορικό εταίρο. Γνωρίζω πλήρω, ε, έχω πλήρη επενδυνόση μάλλον το γεγονότο ότι κάποιοι συνάδελφοι διστάζουν, ιδίω ε, για το αν θα κυρώσει η Σιγκαπούρη τι συμβάσει του ΑΕΛΟ και για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εγώ έχω λάβει εγγυήσει από τον συγκεκριτή David Martin, που έχει κάνει φανταστική δουλειά ω συγγητή, και ο οποίο έχει πιέσει του Σιγκαπουριανού να αναγνωρίσουν πολλέ από τι προτεραιότητε μα, με επιστολή εκ μέρου του Πρωθυπουργού να εκφράζει τι δεσμεύσει και τι υποσχέσει του για τι συμβάσει ΑΕΛΟ και με συμπερίληψη δικτών ε, συγκριτική ε, ε, αξιολόγηση για την περιβαλλοντικά Έχω λάβει όλα αυτά και αυτό δεν είναι μόνο για να σας επενέσω, δεν είναι μόνο για σας κέρδο κέρδος και ένα ένας παραπάνω πόντος Ντέιβιντ, αλλά για ολόκληρη την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Κυρία Γκίλ, ο χρόνος σας τελείωσε. Κύριος Βαλένσης. Βαλένσα. Αύριο θα ψηφίσουμε προκειμένου να διατηρήσουμε το διεθνή, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιριών και να βελτιώσουμε το, το, την ελευθερία του εμπορίου. Με βάση όμως ε, αρχές, τις συγκεκριμένε αρχές που έχουμε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ίσους κανόνες, ίσους όρους και ταυτόχρονα να προστατέψουμε το περιβάλλον. Μερικές φορές είναι δύσκολο για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, αλλά με περηφάνεια θέτουμε διαγραφές προδιαγραφές και πρότυπα στο, στην παγκόσμια σκηνή. Και οι επιχειρήσεις μας μεγαλώνουν. Οι εμπορικές ε, συμφωνίες ε, έχουν οδηγήσει σε αύξηση των ευρωπαϊκών εξαγωγών. Ε, έχουμε το μεγαλύτερο δίκτυο προτιμησιακών συμφωνιών, πάνω από 70 στον κόσμο. Και δημιουργούμε θέσεις εργασία στην Ευρώπη. Και μια ακόμα φορά, οι εμπορικές συμφωνίες με χώρες όπως η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ εφαρμόζονται μία-μία και μας ωφελούν. Θα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ευκαιρίες και στο μέλλον. Αύριο ελπίζω ότι θα υπερψηφίσουμε αυτές τις συμφωνίες. Ευχαριστώ. Dziękuję bardzo. Następny pan wiceprzewodniczący telika poprowadzi dalej. Eh, Οι συμφωνίε αυτέ είναι σημαντικέ για την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν πρέπει να κλειστεί στα σύνορά τη. Αντιθέτω, θα πρέπει να ανοιχτεί στον κόσμο δυναμικά και δραστήρια προκειμένου να ρυθμίσουμε το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Αυτή, αυτές οι συμφωνίες ε, συνεργασίας είναι ένα σημαντικό σημείο φετηρίας για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περιοχή τόσο σημαντική στον κόσμο όπως είναι η Νοτιοτεολική Ασία. Θα αποτελέσει τη βάση για την βελτίωση των διμερών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σιγκαπούρης, θα ενισχύσει τον πολιτικό διάλογο και θα επιτρέψει την καλύτερη συνεργασία σε μια ευρεία σειρά η... Θα αποτελέσει μοντέλο ε, τέτοιων συμφωνιών ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, τα όπλα, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ε, την προστασία του περιβάλλοντος, οι διεθνείς συμφωνία κλπ. Την ενέργεια, τις μεταφορές, όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη, μα ενημέρωσαν ότι έχουμε μείνει 25 λεπτά πίσω από το χρόνο διαγράμμα μα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ο καθένα να σέβεται ακριβώς και να τηρεί το χρόνο ο οποίο του απονέμεται. Δεν θα επιτρέψω μπλε κάρτε. Οπότε μία ακόμα φορά, καλησπέρα σας, ο κ. Πέτρελ έχει το λόγο. Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον David Μάρτιν για την εξαιρετική του έκθεση. Η συνεργασία και η εταιρική σχέση με τη Σιγκαπούρη περιλαμβάνει όχι μόνο την προστασία των επενδύσεων, αλλά μια γενικότερη πολιτική σχέση που θα μας επιτρέψει να συνεργαστούμε πιο εντατικά, πιο στενά και για την προστασία του περιβάλλοντος, για την ασφάλεια, για την ανάπτυξη κλπ. Οι συμφωνίες αυτές ανοίγουν καινούριε ευκαιρίε συνεργασία και στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και άλλους τύπους συνεργασία μεταξύ αυτών και της υγείας. Η συμφωνία αυτή θα μας επιτρέψει να καταπολεμήσουμε μαζί τον καρκίνο και μας ανοίγει τα σύνορα όλης της περιοχής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Η συμφωνία είναι αρκετά ισορροπημένη και εξ όσων γνωρίζω η Σιγκαπούρη έχει δεσμευτεί ότι θα κυρώσει τη συμβάση του το στο μοτρό δυνατόν. Αλλά αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερο σημαντικό είναι η παρακολούθηση των συνεπειών από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Γεγονό είναι ότι η Σιγκαπούρη είναι πάρα πολύ ψηλά όσον αφορά την ε, διαφθορά, δηλαδή θεωρείται μη διαφθαρμένη χώρα, αλλά περιέργως ε, έχει και πολύ ισχυρό τραπεζικό απόρριτο. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν κάποια μέτρα για να ισχύουν αυτά για τα κρατημέλη. Προσφάτως είχαμε ένα πρωτόκολλο αποφυγής διπλής φορολογίας με την ε, Λετωνία για να ενισχυθούν οι αμοιβέ επενδύσεις. Και βεβαίως δεν ξέρουμε το εάν τα ιδιαίτερα δικαιώματα των επενδυτών είναι συμβατά με τα ανθρώπινα και περιβαλλοντικά δικαιώματα. Βεβαίω, πολλά εξαρτώνται εδώ πέρα από την ικανότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να απαιτήσει την εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Σα ευχαριστώ, κύριε Μάμικιν Σδρογεύχη, για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ. Κοιτάξτε, όλη αυτή η υπόθεση ξεκίνησε το 2014 με ένα ερώτημα προς το ΔΕΚ. Λάβαμε τις απαντήσεις το 2017, τώρα έχουμε 2019 και ε, η Ινδονησία, οι Φιλιππίνες και το Βιετνάμ ε, και αυτές ε, περιμένουν την σύναψη νέας συμφωνίας μετά την συμφωνία με την Σιγκαπούρη. Θα ήθελα να πω πως είμαι ιδιαίτερος ικανοποιημένος για την συμφωνία με τον Καναδά. Κατά την άποψή μου η προστασία των επενδύσεων, η αποφυγή διπλής φορολογίας και η έλλειψη δασμών είναι υποφελής για τους εταίρους μας και για εμάς. Πρέπει να μας χαροποιεί να προσθέσω πως οι διαδικασίες που εφαρμόζουμε είναι πολύ δυσκίνητες και θέτουν σε κίνδυνο τους δεσμούς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να δούμε πώς μπορούν να γίνουν ε, πιο γρήγοροι. Σας ευχαριστώ. Μπουσό για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω την Συμφωνία Εταιρικής ε, Σχέσης και συγχαίρω τις διαπραγματευτικές ομάδες. Η Σιγκαπούρη είναι εδώ και καιρό ένας αξιόπιστος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φιλοξενεί χιλιάδε ευρωπαϊκές εταιρείες και βεβαίως ε, έχει τις ίδιες αξίες με εμάς για μια ελεύθερη και ανταγωνιστική οικονομία και κράτος δικαίου. Ιδρυτικό μέλος του ΑΖΙΑΝ, μεγάλος κόμβος της ε, περιοχής και εγώ θεωρώ ότι ε, η σχέση αυτή έχει στη βαρύ γεωστρατηγική βάση για την μελλοντική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Αζίαν. Η συμφωνία αυτή θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες εξαγωγής ε, για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και έτσι θα δώσει μια όθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία 550 εκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα 10 χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία και the Λοιπόν, ε, κλείνει εδώ ο κατάλογος. Πρώτος στο λόγο έχει ο κύριος Πόσπισιλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω τον θαυμασμό μου για εσάς ε, κυρία Επίτροπε επειδή οριστικοποιήσατε αυτήν την ε, συμφωνία. Θα πρέπει να προωθούμε τις αρχές του ελευθέρου εμπορίου ε, σε αντίθεση με την τωρινή Αμερικανική κυβέρνηση. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι στο μέλλον. Πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι σε τέτοιες ε, συμφωνίες ε, και να μειωθεί ο χρόνος της διαπραγμάτευσης. Μου πέρασε σχεδόν 10 χρόνια βεβαίως. είχε εμπλακεί και το δικαστήριο, αλλά ας σκεφτούμε το τι πρέπει να κάνουμε για να μπορούμε να υπογράφουμε τέτοιες συμφωνίες πιο γρήγορα. Ελπίζω λοιπόν σιγά σιγά να υπογράψουμε διμερείς συμφωνίες με, ολόκληρες τις, με όλες τις χώρες του ΑΖΙΑΝ. Ε, το ελευθερεμπόριο πρέπει να είναι η ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στον κόσμο. Πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω πως ε, πιστεύω στο ελεύθερο εμπόριο που θα βασίζεται όμως σε κάποιες κοινέ αξίες και έχουμε κάποιες ε, κοινέ αξίες ε, με την Σιγκαπούρη δηλαδή τις φιλελεύθερες τάσεις, το κράτος δικαίου κτλ. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τους ηγητές και τις διαπραγματευτικές ομάδες. Νομίζω ότι βρήκαμε μια ισορροπημένη συμφωνία που αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τι εταιρείε μα τους πολίτε μας, ε, τα θεσμικά όργανα. Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλη συμφωνία θα μπορούσαμε να επιτύχουμε. Υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις, αλλά δεν υπάρχει κάποια άλλη συμφωνία. Απλά θα χάσουμε χρόνο. Οπότε είμαι υπέρ αυτή τη συμφωνία. και σα ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε των σχέσεων με την ε, Σιγκαπούρη είναι θετική, ανοίγει ένα σημαντικό τομέα εμπορίου και μας δίνει δυνατότητα να με, βελτιώσουμε τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή. Και βεβαίως ε, υπάρχουν ε, οι κίνδυνοι που είχαμε δει και στην περίπτωση της TTIP, μια μορφή του ISDS, ένα διεθνές ε, δίκαιο το οποίο εγγυάται έναν ιδιαίτερο μηχανισμό επίλυσης διαφορών των επενδυτών με, ξένες, ε, με ξένα κράτη. πρόκειται για ένα μεγάλο λάθος. Ανταυτού θα πρέπει να προχωρήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα υποχρεώνει τις ε, επιχειρήσεις να πληρώνουν για τις παραβιάσεις δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος. Λοιπόν, η συμφωνία αυτή είναι η πρώτη και θα αποτελέσει υπόδειγμα για τις συμφωνίες με Κίνα και με άλλες μεγάλες οικονομίες. Σας ευχαριστώ κύριος Μαριές για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Σιγκαπούρης οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση του εμπορίου και αυτό σημαίνει φυσικά αθρώες εισαγωγές φθηνών προϊόντων από την Σιγκαπούρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι η Σιγκαπούρη στην πράξη είναι το προγεφύρωμα τη Κίνα. Εκεί εισάγονται με τον ΑΒ τρόπο κινέζικα προϊόντα τα οποία εν συνεχεία θα εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και όσα κατασκευάζονται στη Σιγκαπούρη, εκεί ξέρουμε όλοι ότι δεν τηρείται η εργατική νομοθεσία. Έχουμε ένα κλασικό μισθολογικό ντάμπινγκ. Έχουμε επί τη ουσία μια διαδικασία η οποία παραβιάζει οποιαδήποτε έννοια δικαίου εμπορίου. Είναι μια περιοχή η Σιγκαπούρη που αξιοποιείται από του μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της ευρωπαϊκής ένωσης και άλλων χωρών για τη δημιουργία υπερκερδών. είμαι ενάντια φυσικά και στην λογική του isds που υπάρχει που επί του πρακτέου προστατεύει τους επενδυτές εις βάρος των κρατών και τέλος η ευρωπαϊκή ένωση φαίνεται ότι έχει ξεχάσει ότι στη σιγκαπούρη δεν τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζεται το κράτος δικαίου παραβιάζεται κάθε δημοκρατική έκφραση και ισχύει ακόμη That Σας ευχαριστώ. Τελειώσαμε έτσι με τον ε, κατάλογο. Κυρία Επίτροπε, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να απαντήσω μερικές ερωτήσεις. Το ε, κρατικό χρέος εξαιρείται ε, είναι σαφές ότι εξαιρείται το κρατικό χρέος από, και η αναδιάρθρωσή του από την προστασία των επενδύσεων. Ε, ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών, ο ISDS, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει πλέον. Τον έχουμε αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό χάρη στην δική σας παρέμβαση και πιέσεις με ένα, από ένα νέο, μοντέρνο, σύγχρονο σύστημα το οποίο ο Γενικός Αγγελέας ε, ανέφερε ότι κήρυξε απόλυτα συμμορφούμενο με την ε, ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ε, πλήρης διαφάνεια, διοντολογικός κώδικας, είναι σαφές ποιος μπορεί να προσφέρει και για ποιο λόγο και αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να ρυθμίζουν τις αγορές τους και την οικονομία τους. Ε, δεν, η Σιγκαπούρη δεν αποτελεί φορολογικό παράγοντα, ε, παράδεισο. Ε, είναι προφανές ότι ε, έχουμε δουλειά να κάνουμε για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Ε, η Σιγκαπούρη θα δημιουργήσει ένα μητρό και οι ευρωπαϊκές ε, χώρες θα μπορέσουν να ζητήσουν τη συμπερίληψη των 196 προϊόντων τα οποία είχαμε ήδη απαριθμίσει. Είναι αλήθεια ότι η Σιγκαπούρη θα πρέπει ακόμα να επικυρώσει τρεις συμβάσεις του ILO αλλά γίνεται ήδη πολύ σοβαρή δουλειά στην εσωτερικά στην κυβέρνηση ε, της Σιγκαπούρης σε συνεργασία με τον ΆΕΛΟ, έτσι ώστε πράγματι να ε, προσαρμοστεί η νομοθεσία της Σιγκαπούρης και να ευθυγραμμιστεί με αυτές τις συμβάσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να επικυρωθούν. Όπως είπατε και εσείς, η κυβέρνηση Σιγκαπούρης έστειλε μια επιστολή για την διαδικασία αυτή. Αν υπερψηφίσετε αύριο με μεγάλη πλειοψηφία, τι συμφωνίε αυτέ και ελπίζω θα το κάνετε θα ψηφίσετε υπέρ μια φιλόδοξη συμφωνία ελεύθερων, ε, ελεύθερων πορείου που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για πολλέ άλλε μελλοντικέ συμφωνίε με τι χώρε τη περιοχή αυτή της Ασίας. Είμαστε υπέρ τη Συμφωνία Προστασία των Επενδύσεων που ακολουθεί την προσέγγιση την οποία εσεί βοηθήσατε να αναπτυχθεί. Θα βοηθήσετε με αυτόν τον τρόπο ε, την τοποθέτηση της ευρύτερης συνεργασίας σε ένα συγκεκριμένο σαφές και σταθερό πλαίσιο σε θέματα όπως ασφάλεια, ε, έρευνα, μέσω της ε, εταιρικής συμφωνίας και θα είναι και η πρώτη συμφωνία την οποία θα εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την καινούρια σύγχρονη ε, αρχιτεκτονική. Με αυτόν τον τρόπο διευρύνουμε τον κύκλο των φίλων μας σε χώρες οι οποίες πιστεύουν στην πολυμερή προσέγγιση, που πιστεύουν στους παγκόσμιους κανόνες χώρες οι οποίες πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα να υπογράφουμε, να συνάπτουμε εμπορικέ συμφωνίε που θα είναι ωφέλιμε και προς, για τι δύο πλευρέ. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ελέγξουμε την παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Σα ευχαριστούμε. Ε, και αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να επενέσω το έργο σας και εγώ. Ένας από τους δύο εισηγητές ε, πήρε ε, όλο το χρόνο που χρειαζόταν στην αρχή, που είχε στην αρχή, οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάρτιν. Η κυρία Μάλιστρο μου απάντησε πολλές από τις ερωτήσεις, αλλά κοιτώ εδώ γύρω και δεν βλέπω κανέναν από αυτούς που επέκριναν τη συμφωνία να είναι εδώ παρόν. Οπότε σε ποιον να απαντήσω. Να, να πω όμω, να επαναλάβω ότι σε ό,τι αφορά την ε, Συμφωνία Ελεύθερων Ανταλλαγών, είναι καλή για την απασχόληση, για τι επενδύσει. Ε, σε ό,τι δεν αφορά τι επενδύσει, είναι η πιο σύγχρονη συμφωνία που έχουμε μέχρι τώρα και θα συμφωνήσω με την Επίτροπο σε αυτό που είπε. Προσπαθούμε να διαβρύνουμε τι σχέσει μα με χώρε οι οποίε σκέπτονται με τον ίδιο τρόπο που σκεπτόμαστε εμείς. Κάποιες άλλες χώρες προτιμούν τον νόμο της ζούγκλας. Εμεί προτιμούμε κοινού πολυμερείς κανόνες. Ευχαριστώ. Άρα καταλαβαίνω ότι οι συνάδελφοι που δεν είχαν αρκετό χρονομιλία ε, θα πίστηκαν φαντάζομαι ε, στη διάρκεια των όσων άκουσαν. Ευχαριστώ συνάδελφοι, κοινή συζήτηση ολοκληρώθηκε, η ψηφοφορία είναι αύριο και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα που είναι η προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η υποβάθμιση τα δικαιώματα των γυναικών και στη ισότητα των φίλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο συντάκτης είναι ο κύριος Πιμέντα Λόπες. Θα του δώσω το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, επιτρέψτε μου πάνω απ' όλα να σας πω ότι ε, είχαμε πολύ καλή συνεργασία με όλους τους συναδέλφους που βοήθησαν στη σύνταξη της προφορικής αυτερότητας και του ψηφίσματος. Είναι σαφές ότι η υποφάθμιση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φίλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει να δείξουμε καμία ευλεψία και αμέλεια. Τα τελευταία δέκα χρόνια τα κοινωνικά εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα των γυναικών υποβαθμίστηκαν σοβαρά. Οι πολιτικές της δεξιάς ε, με, ε, υπό την αιγίδα μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως επιβλήθηκαν οδήγησαν σε επισφάλεια των εργασιακών σε, μάλλον ε, επισφάλεια στι εργασιακέ σχέσει, την υποβάθμιση των εργασιακών συμβάσεων, κατοίκη μεταχείριση ει βάρο των γυναικών. Και οι κοινωνικέ ε, αποκρίσει, η κοινωνική κάλυψη, η προσφορά δημοσίων υπηρεσιών ε, περιορίστηκαν για τη φροντίδα, την υποστήριξη, τι περιπτώσει αρρώστια, γυρατιών ε, την ανάληψη ευθυνών από τα κράτη ε, που δεν μπορούν πλέον να καλύψουν τέτοιου είδου περιπτώσει. Όλα αυτά δημιούργησαν καταστάσει που αποκλείουν τις γυναίκες από την αγορά εργασίας. Η μητρότητα, όπως ε, καθορίζεται από το δίκαιο, ε, είναι μια τεράστια πίεση εις βάρος των εργαζομένων για να καταλήψουν τα δικαιώματά τους ή γίνονται επισφαλείς οι εργασιακές τους σχέσεις. Η δημόσια προσφορά υγειονομικής περίθαλψης ή ε, ο περιορισμός των υπηρεσιών για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία περιορίζουν τα δικαιώματα των γυναικών. Είναι γνωστά και απαράδεκτα όσα γίνονται με τις απόπειρε να μην υπάρχει το δικαίωμα στην οικειοθελή διακοπή της κοίησης και να μην προσφέρονται απαραίτητες υπηρεσίες για την απορροφική υγεία. Τα παγκόσμια επίπεδα φτώχεια και ενεργεία που πλήττουν κυρίω τι γυναίκε παραμένουν σε ποσοστά που δεν μπορούν πλέον να συνεχιστούν. Ε, το χάσμα μυστολογικό και συνταξιδοτικό μεταξύ άνδρων και γυναικών παραμένει απαράδεκτο. Επίση, αυξάνονται τα φαινόμενα βία κατά των γυναικών. Βλέπουμε ότι την ίδια περίοδο αυξάνονται τα φαινόμενα αυτά. Και αυτό ε, δείχνει ότι υπάρχει υποβάθμιση των κοινωνικονομικών ε, συνθήκων ε, για όλο τον πληθυσμό και για τις γυναίκες. Ήταν δεκάδες οι γυναίκες και τα παιδιά που ήταν θύματα οικογενειακής βία από την αρχή της χρονιά στη χώρα μου. Αυτά δείχνουν ότι η βία διωγγώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω οι μορφέ βία συμπεριφορά κατά των γυναικών, είτε ενδογενειακή, είτε σεξουαλική, είτε εργασιακή ε, και διακριτική μεταχείριση του φύλου, είτε σε ε, ε, επίπεδο θεσμικό. Θα πρέπει η βία να μην καλύπτεται από τον νόμο, είτε διεθνώ είτε εθνικό. Πρέπει να εγκριθεί η σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Βήματα απαραίτητα ε, και αναγκαία. Ε, αλλά δεν αρκεί η παγίωση ορισμένων δικαιωμάτων στο δίκαιο. Θα πρέπει να υπάρχει και πολιτική που θα υποστηρίξει την ισότητα των φίλων, που θα καταπολεμήσει κάθε μορφή και έκφραση βία. Το αποτέλεσμα τη πολιτική δράση, τη καταπολέμηση και τη εκρίζωση τη βία κατά των γυναικών, στι πολλαπλέ εκφράσει τη, είναι αλληλένδετο με την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών γυναικών, όπω τα εκφράζονται στο δίκαιο και στον καθημερινό επαγγελματικό και οικογενειακό βίο. Θα πρέπει να, να προσφερθεί προστασία στα θύματα, κοινωνική υποστήριξη, πρόσβαση στη δικαιοσύνη, εκδίκαση των υποθέσεων, ε, στήριξη στην ψυχολογική ε, υγεία του, ε, αποκατάσταση, οικονομική ανεξαρτησία και στην πράξη να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη του, την ασφάλεια ότι ο νόμο πραγματικά προστατεύει τι γυναίκε θύματα τη βία στα διάφορα στάδια εξέλιξη τη ζωή του. Η οικονομική και κοινωνική χειραφέτηση των γυναικών είναι καθοριστική σημασία για τη δημιουργία τη ισότητα και την καταπολέμηση όλων των μορφών βία και πρέπει να βρεθούν ε, στο χώρο εργασίας σε κεντρικό ρόλο για να αντιμετωπίσουν τις ανισότητες. Θα πρέπει η ανεργία και η επισπάλεια των θέσεων εργασίας, η μισθολογική διάκριση ή το χάσμα μισθού ανδρών γυναικών, η συμμετοχή των γυναικών ε, σε συνθήκε ισότητας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής δράσης, η, τα ισότιμα δικαιώματα για τους εργαζομένους, η άδεια μετρότητας και πατρότητα, ε, η κοινωνική διάσταση, η στη δυναμική περίθαλψη, στη σεξουαλική αναπαραγωγική υγεία, οι εγκαταστάσει που θα προσφέρει βοήθεια στα παιδιά, του νέου, του ηλικιωμένου, στα θύματα τη βία, η πρόσβαση όλων στην ε, ε, προστασία τη υγεία και την προστασία τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, ε, προστασία των γυναικών που είναι θύματα δικτύων πορνεία ή εμπορία που τι έχουν οδηγήσει πάλι στο ίδιο αποτέλεσμα, πρέπει να οργανωθούν. Πρέπει όλα τα κράτη να καταπολεμήσουν τα φαινόμενα αυτά, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να καταλάβουν ότι είναι μια στιγμή στην οποία πρέπει οπωσδήποτε να αναλυφθεί δράση για την παγίωση της ισότητας ως ενός παράγοντα που θα ισχύει σε όλη μας την νομοθεσία. Ευχαριστούμε. η κυρία Γιούροβα τώρα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτές, η Ευρώπη αντιμετωπίζει διάφορες ε, λαϊκιστικές ε, κινήσεις, οι οποίες επίσης εκφράζονται με τρόπο σεξιστικό και ρατσιστικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την στήριξη της κυρίας Μογκερίνη έχει θέσει το θέμα του φύλου στο επίκεντρο της εξωτερικής της ε, δράσης. Η στρατηγική για την ισότητα το 2016-2019 απετέλεσε το πλαίσιο της ε, προώθησης της ισότητας των φύλων το 2019 κάνουμε έναν απολογισμό της ε, προόδου βλέπουμε ποια είναι τα κενά και εξετάζουμε τις προτεραιότητες μας για το μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό οι απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ σημαντικές. Επίσης ε, καλωσορίζω την ε, συμφωνία που επετεύχθη για την πρόταση ισορροπίας οικογενειακής και προσωπικής ζωής για να μπορέσουν έτσι οι να τις συμβιβάσουν. Το Νοέμβριο του 2017 η Κομισιόν έκανε ένα σχέδιο δράσης για να αντιμετωπίσει το μισθολογικό χάσμα και είχαμε 20 συγκεκριμένες δράσεις, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν εφαρμοστεί και οι υπόλοιπες θα ολοκληρωθούν φέτος. Αξιόπιστα δεδομένα επίσης έχουμε καλή για να παρατηρούμε τις τάσεις στην ισότητα των φύλων. Γι' αυτό η Eurostat αυτή τη στιγμή αναπτύσσει μια πανευρωπαϊκή έρευνα για την βία για να έχουμε ενημερές, ενημερά στατιστικά στοιχεία με βάση τον σχετικό κανονισμό του 2014. Η εξάλληψη της βίας με βάση το φύλλο είναι βασική προτεραιότητα της ε, Κομισιόν. Μόλις ολοκληρώσαμε ένα δεύτερο έτος στοχευμένων δράσεων και ενημέρωσης και συνεχίζουμε να προωθούμε την υπογραφή της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι σήμερα 20 κράτη-μέλη έχουν κυρώσει αυτή την σύμβαση, αλλά όπως ξέρετε υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις σε άλλες χώρες. Η πολιτική και η δημόσια συζήτηση ακριβώς δείχνει το κλίμα το οποίο αναφέρει η ερώτηση. Έχουμε παραπλανητικά επιχειρήματα για την σύμβαση αυτή, τα οποία χρησιμοποιούνται στην ε, δημόσια συζήτηση. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και να εξηγήσουμε ότι ο μόνος στόχος της σύμβασης αυτής ε, είναι να προλάβει και να καταπολεμήσει τη βία βάρος των γυναικών ε, και γενικώ την ενδοοικογενειακή βία. Η κατάσταση αυτή παραλύει κάποια κράτη-μέλη και έτσι δεν προχωρούν στην ε, κύρωση και δεν μπορεί να ενταχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην συνθήκη και ο χρόνος τελειώνει αν είναι να γίνει κάτι τέτοιο πριν λήξει η θητεία του Κοινοβουλίου. Βεβαίω αυτό έχει σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την εξωτερική μας ε, δράση. Χαίρομαι για το ότι το Κοινοβούλιο καλωσορίζει την πρόοδο στους τομείς ε, διεθνούς συνεργασίας και στο σχέδιο δράσης για το φύλλο. Εκεί πέρα εστιάζουμε σε ζητήματα κεραιότητας ε, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και την κατάργηση της βίας με βάση το φύλλο το Συμβούλιο καλωσόρισε τη νέα φιλόδοξη στρατηγική για τις γυναίκες και την ειρήνη που ρητά συνδυάζει εσωτερική και εξωτερική πολιτική και ζητάει την ανάλυση και αντίδραση στα ε, ζητήματα αυτά, δηλαδή τις ανισότητες, ε, την βία και την σύγκρουση. Τέλος, ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Γι' αυτό ακριβώς τον Σεπτέμβριο του 2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τον ΟΗΕ ξεκίνησε μια πρωτοβουλία με στόχο να απαλληφθούν όλες οι μορφές βίας κατά γυναικών και κοριτσιών παγκοσμίω. Και βεβαίως με 500 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση σκοπεύουμε η πρωτοβουλία αυτή να αλλάξει τις ζωές γυναικών και κοριτσιών σε ολόκληρο τον κόσμο, ειδικά για τους νέους και για όσους ζουν σε καταστάσεις όπου είναι περιθωριοποιημένοι. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και βασίζομαι και στην δέσμευση Κοινοβουλίου και Κομίσιον. Σας ευχαριστώ. Παίρναμε τώρα στους ομιλητές ε, εξ των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Πιετικάνη για το ΕΛΚ. Οι κοινωνίες μας, ε, στις κοινωνίες που είναι ανοιχτές, ε, Συνήθω οι γυναίκες τα πάνε καλά. Και όταν οι γυναίκες τα πάνε καλά, τα πάνε καλά και οι κοινωνίες. Γι' αυτό το λόγο, η θέση των γυναικών είναι σαν το καναρίνι στα ορυχεία. Γιατί προειδοποιεί για, την, για το τι θα επικρατήσει. Οπότε όταν οι γυναίκες υποφέρουν, αυτό δείχνει ότι οι κοινωνίες οδηγούνται προς τον περιορισμό της δημοκρατίας του ε, κράτους της ε, ε, ε, ευημερίας και της αλληλεγγύης. Και αυτοί που υφίστανται διακρίσεις δεν είναι μόνο γυναίκες βέβαια, αλλά τουλάχιστον οι, οι μισές είναι γυναίκε και μάλιστα δεν είναι μόνο εργαζόμενε, είναι και επιχειρηματίε, είναι και μετανάστε, είναι και μειονότητε κλπ. Και είδαμε αυτή την εναντίωση και την οπισθοδρόμηση τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα, τα δικαιώματα των γυναικών συμπεριλαμβάνουν τα δικαιώματα της αναπαραγωγής και τα σεξουαλικά δικαιώματα και αποτελούν τμήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οπότε η οπισθοδρόμηση στα δικαιώματα των γυναικών αποτελεί απιστοδρόμηση στα ανθρώπινα δικαιώματα γενικά. Ευχαριστώ. Κυρία Γκαρθία, Γκαρθία Πέρεθ, για δύο λεπτά, για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Μιλάμε για την οπισθοδρόμηση των δικαιωμάτων γυναικών στην Ευρώπη. Το 2014, πριν από πέντε χρόνια, συζητούσαμε εδώ ακριβώς τα δικαιώματα, τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και τα δικαιώματα σεξουαλική υγεία των γυναικών. Και έλεγα ότι να, δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε οι κόρε μα να έχουν λιγότερα δικαιώματα από ότι οι μητέρε μα. Ε, αυτή τη στιγμή ζούμε αυτή την απειλή. Η Πολωνία με τον νόμο περί αμβλώσεων, η Ουγγαρία που ε, καταργεί τις, ε, ε, τις σπουδές, ε, γυναικές σπουδές στα πανεπιστήμια της, η Βουλγαρία που θέλει να βγει από τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης κλπ. Και ε, το ε, συντηρητικό κόμμα στην ε, Ισπανία λέει ότι για να γλιτώσει το σύστημα το ε, κοινωνικής ασφάλισης στην Ισπανία θα πρέπει εμείς να κάνουμε περισσότερα παιδιά. Αυτό είναι μεγάλη οπισθοδρόμηση ως επιχείρημα. Οι γυναίκες έχουν χαμηλότερου μισθού, χαμηλότερε συντάξει, δυσκολεύονται περισσότερο στο να ενταχθούν στην αγορά εργασία. Φροντίζουν τα, άτομα, τα εξαρτώμενα άτομα τη οικογένειά του. Και κάθε μέρα δολοφονούνται γυναίκε από ανδρική βία. Είναι, είμαστε θύματα σεξουαλικής βίας και εμπορίου ανθρώπων. Οι γυναίκες, πολλές φορές μάλιστα, έχουμε, φοβόμαστε να γυρίσουμε και μόνοι μας στο σπίτι. Δεν είναι δυνατόν να παραμείνουμε ε, άμυρες ε, ε, και αδιάφορες σε αυτή την κατάσταση. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι, και υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Πρέπει να κινητοποιήσουμε τις γυναίκες να συμμετάσχουν στην απεργία της 8 Μαρτίου. Θα πρέπει να γεμίσουμε τους δρόμους και να διεκδικήσουμε ισότητα. Γιατί το θέμα αυτό δεν αφορά τις γυναίκες. Είναι ένα θέμα ε, ε, είναι, έχει σχέση με τον αγώνα για μια Ευρώπη των γυναικών που δεν υποχωρούν ε, και δεν παραδίδονται. Ευχαριστώ. No, but uh, we are not taking cards. announced uh, uh, Όχι, όχι. Συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε με την διαδικασία και HDI, αλλά δεν θα επιτρέψω μπλε κάρτες γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει 25 λεπτά. Ζητώ συγγνώμη. Κυρία Βυσνιεύσκα, για ένα μισή λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, είναι προφανές ότι είμαι υπέρ της ισότητας των γυναικών. Αλλά δεν συμφωνώ με κάποιες υποθέσεις εδώ πέρα και τα βασικά στοιχεία αυτού του ψηφίσματος. Πρώτα απ' όλα γιατί ε, στόχο έχει να περιορίσει την ελευθερία λόγου. Με το να ε, ε, μην μπορεί κανείς να ασκήσει κριτική στην σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και λέει ότι μητρότητα, μα λέτε, θα εμποδίσει τις γυναίκες στην επαγγελματική του αδειοδρομία. Δεν συμφωνώ με αυτό. Και επιπλέον... Ε, Βλέπουμε ότι γίνεται μία έκκληση σε σχέση με κάποια στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι αποτελούν εδώ πέρα παραπληροφόρηση. Λοιπόν, δεν συμφωνώ με αυτό το οποίο λέγεται στο ψήφισμα αυτό όσον αφορά τις αμβλώσεις. Ότι τα όσα ισχύουν για τις αμβλώσεις αντιστοιχούν ουσιαστικά σε μία αποδυνάμωση των δικαιωμάτων των γυναικών. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα άλλο ψήφισμα. Ένα ψήφισμα το οποίο εστιάζεται περισσότερο στο μισθολογικό χάσμα, το οποίο εστιάζεται περισσότερο στην, στον ακροτεριασμό των γεννητικών οργάνων. Ένα ψήφισμα το οποίο αναφέρεται περισσότερο στους αναγκαστικούς γάμους. Ένα ψήφισμα το οποίο να προωθεί περισσότερο τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή. Η κυρία Μινάρτο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, να ευχαριστήσω καταρχάς τον εισηγητή και τους σκιώδη εισηγητές για την πολύ επικοδομητική συνεργασία που είχαμε για το ψήφισμα αυτό. Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο διακριτική μεταχείριση και δεν συμμετέχουν ισότιμα στην πολιτική, οικονομική κοινωνική ζωή και δέχονται επίσης πολλές φορές κακοποίηση τόσο ενδοκογενειακή όσο και στον χώρο εργασία. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια εναντίωση αυτή τη στιγμή στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φίλων. Τα επιτεύγματα των τελευταίων δεκαετιών είναι ακόμα εύθραστα και θα πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν πολλέ πολιτικέ και θρησκευτικέ ομάδε, οι δύο θρησκευτικέ ομάδε που χρησιμοποιούν πολύ συχνά πολιτιστικά στοιχεία ακριβώ για να στραφούν κατά των δικαιωμάτων των γυναικών. Και αναφέρουμε αυτή τη στιγμή και σε κάποιε ομάδε οι οποίε αρνούνται στι γυναίκε το δικαίωμα στην άμβλωση ή το δικαίωμα στην, στον ισότιμο μισθό. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία συνάδουν στην εναντίωση αυτή στα δικαιώματα των γυναικών. Στο ψήφισμα λοιπόν αυτό ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε πραγματικέ πράξει. Καλούμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα επιμέρου κράτη-μέλη να επιταχύνουν την εφαρμογή των δικαιωμάτων των γυναικών, να επιταχύνουν την αποτελεσματική λειτουργία όλων των μέσων που προστατεύουν τα δικαιώματα των γυναικών και επίση ζητούμε να γίνουν περισσότερε επενδύσει στου οργανισμού εκείνους που προωθούν τα δικαιώματα των γυναικών. Είναι πολύ σημαντικό εθνικοί αλλά και περιφερειακοί προπολογισμοί να προβλέπουν συγκεκριμένα κονδύλια προκειμένου να προασπίζουν τα δικαιώματα των γυναικών. Και αυτό θα πρέπει να αποτελεί θέμα συζήτησης ε, σε όλες τις συζητήσεις που γίνονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό το έργο των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών. Πρώτα κυρίως για γυναίκες, αλλά γενικότερα για πολίτες μας, οι οποίοι δέχονται πάρα πολλές επιθέσεις, μόνο και μόνο επειδή υποστηρίζουν τα δικαιώματα των γυναικών. Από την Ενωτική Αριστερά, κύριε Πιόρκ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε είναι κεντρικό στοιχείο της δημοκρατίας, οι γυναίκες. Και αυτό ε, θα πρέπει να είναι αυτονόητο το 2019 για τα γυναικεία δικαιώματα. Βλέπουμε όμως ότι τώρα υφίστανται επιθέσεις και ε, οπισθοδρόμηση υποχωρούν τα ε, γυναικεία δικαιώματα. Η δεξιά και η ακροδεξιά ε, απειλούν τα γυναικεία δικαιώματα. Υπάρχουν και προβλήματα υλικά. Η ανεργία, το μειωμένο εισόδημα, η μειωμένη πρόσβαση ε, σε δημόσιες υπηρεσίες και ε, οι ακτιβίστριες δέχονται επιθέσεις. Δεν είναι νομοτελειακό το να προχωρούν τα γυναικεία δικαιώματα. Αυτό το έλεγε η μητέρα μου πάντα. Δεν είναι αυτονόητο ότι όσο προχωράει ο καιρός τα δικαιώματα ε, θα κατακτώνται. Δεν μπορούμε να ε, επιτρέψουμε αυτή την οπισθοδρόμηση. Θα πρέπει να απαιτούμε να προχωρούμε. Αυτή η φεμινιστική πάλι και μάχη δεν πρόκειται ποτέ να ε, συνθηκολογήσει. Δεν θα δεχτούμε από κανέναν συντηρητικό τέτοια φαινόμενα. Η κυρία Ράιντκε, στη Βουλγαρία ε, ο κόσμος ε, ε, μαθαίνει ψευδείς ειδήσει για τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Σε άλλη χώρα, στην Πολωνία, λένε ότι η μόνη φυσική μορφή αντισύλληψης είναι ε, ο υπολογισμός της οφλακυρωξία. Ε, υπάρχουν τεράστιε επιθέσει παντού στα γυναικεία δικαιώματα. Ε, τα επιτεύγματα και οι κατακτήσεις ε, πλήττονται κυρίως στις γυναίκες. Ο έλεγχος του σώματος των γυναικών είναι πρώτη προτεραιότητα χριστιανικών φονταμεταλιστών και νεοσυντηρητικών. Υπάρχει και λασπολογία τεράστια ε, κατά τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και υποδάβληση μίσους κατά τον ΛΟΑΔ και με χρήματα, όχι μόνο με λόγια, από την Ηνωμένε Πολιτείε και από την ε, Ρωσία οι ολιγάρχες για να γυρίσει πίσω το ρολόι. Εμείς τι κάναμε, αδρανίσαμε πάρα πολύ καιρό και τώρα θα πρέπει να σταματήσουν αυτά ανοίγουμε το στόμα μας και αντιστεκόμαστε κατά των φαινομένων αυτών και όσων θέλουν να φημώσουν τις γυναίκες. Και όποιος ε, θέλει να επαναφέρει ρατσιστική και πατριαρχική υποτίθεται φυσική τάξη θα μας βρει απέναντί του. Και πού ξεκινάμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Ο πρόεδρος Αντώνιο Ταγιάννη ε, είπε ότι θα πάει στη Βερόνα σε μια συνεδρίαση αντιδραστικών ομάδων. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν αισθάνεται ε, ε, ότι αγωνίζονται για τα ε, δικαιώματα θα πρέπει να ματαιώσει τη συμμετοχή του εκεί. Ο Πρόεδρος, έχουμε καθυστερήσει πολύ και θα πρέπει να σεβόμαστε το χρόνο. Ο κύριος Σόσνης, για ένα λεπτό, μη εγγεγραμμένος. Ε, ανησυχείτε για τα γυναικεία δικαιώματα. μα τι είναι αυτά που λέτε. Τι είναι αυτές οι ανοησίες για τη διάκριξη και την έλλειψη ισότητας. Αυτό που υπάρχει είναι ότι δεν σας υποστηρίζουν στα λεγόμενά σας, διότι η κοινωνία μας ε, έχει κατακλειστεί από προπαγάνδα για την πάλη των φίλων, για τον πόλεμο των φίλων. Δεν είναι τα, ε, τα ίδια τα χρώματα, σώματα, το χ και το ψ, ε, το χ και το ύψιλον μάλλον. Ε, αυτές τις ανοησίες που λέτε εδώ, πρέπει να ακούτε τι λέτε. Δεν πιάνουν τόπο, δεν σας ακούει ο κόσμος. Ε, τα αντίθετα ισχύουν. Ε, εάν δεν δικαιώνεστε, σημαίνει ότι είναι λάθος η απόψη σας. Και πού καταλήγουν οι φιμενιστές και οι μία από τα ίδια. Και άλλα ψηφίσματα και άλλες προφορικές ερωτήσεις και άλλες προσφυγές και συνεχίζεται να εκνευρίζεται τον κόσμο άσκοπα. Η κυρία Κουσλόφσκα Ράγεβιτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Επίτροπα κυρίες και κύριοι. Τα δικαιώματα των γυναικών και στο παρελθόν αλλά και τώρα ανήκουν στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν υπάρχει ε, κάτι περισσότερο σε πολιτική οργάνωση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, με την άνοδο της ακροδεξιάς έχουμε αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις και προς τα δικαιώματα των γυναικών. Ε, σε ό,τι αφορά την ε, αναπαραγωγική υγεία των γυναικών. Χρειάζονται ε, συνταγές ε, για να πάρουν τα φαρμακά τους. Ε, υπάρχει, υπάρχουν περιορισμοί στη χρηματοδότηση της γυναικείας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που τελικά μα κάνουν να απορούμε κατά πόσο ζούμε στον 21ο αιώνα. Έχει έρθει η ώρα, κυρία Επίτροπε, λοιπόν, να εξετάσουμε τυχόν δυνατότητε παρέμβαση και αξιοποίηση όλων των δυνατών ευκαιριών που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι δυσμένε επιπτώσει. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε παρά τι ε, νομικέ πράξει, συστάσει και στρατηγικέ που έχουν υιοθετηθεί κατά το παρελθόν, στην πράξη είμαστε στα μισά του δρόμου προ την ε, ισότητα μεταξύ των φύλων. Αυτή τη στιγμή η πρόοδο είναι εξαιρετικά αργή και σε κάποιου ε, τομεί τα δικαιώματα των γυναικών όλα είναι και υποβαθμίζονται. Πρώτα απ' όλα, Μέχρι τώρα δεν έχουμε καταφέρει να εξαλείψουμε την γία κατά, τη βία κατά των γυναικών, που είναι μία από τι ε, μείζονε παραβιάσει και καταπατήσει ε, ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμα υιοθετήσει και κυρώσει την Συνδίκη τη Κωνσταντινούπολη. Αυτό συμβαίνει ότι έχουν εξαλείψει την βία κατά των γυναικών ή την έλλειψη πολιτική βούληση για την κύρωση αυτών των νομικών πράξεων. Ακόμα δεν έχουμε καλύψει το χάσμα στι ε, αμοιβέ μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στι συντάξει το χάσμα είναι 40%. Δεν υπάρχει πρόοδο ε, στην λήψη αποφάσεων και στην πολιτική, γιατί οι γυναίκε ακόμα μάχονται να ε, διασφαλίσουν τα ίδια δικαιώματα με του άντρε στον πολιτικό στίβο. Στη δική μου κυβέρνηση τη Λιθουανία δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα. Τόμασιτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, η διάκριση κατά των γυναικών σε πολλούς τομείς θα πρέπει να καταπολεμηθεί και να καταπολεμάται παντού και πάντα. Οι γυναίκες ε, που ε, υφίστανται διακρίσεις μόνο και μόνο εξαιτία του φίλου τους είναι ένα φαινόμενο που προκύπτει από το πολιτικό μας περιβάλλον Κάποιες ε, κοινωνικές ομάδες έχουν ε, ξεκάθαρη στάση και θα πρέπει κάποιος να έχει τη δυνατότητα να διαλέξει τη ζωή που θέλει να ε, διάγει. Όμως βλέπουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει. Πρόκειται για απλό σεβασμό προς τις γυναίκες που επιλέγουν να ζουν διαφορετικά. Σεβασμό προς το δικαίωμα στη ζωή. Αυτό δεν είναι ε, δυσμενής επίπτωση ε, προς ε, τις γυναίκες και εναντίωση στα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ. Είπα από την αρχή όταν ξεκίνησαν τις συνεδρίες ότι είχαμε, έχουμε μεγάλη καθυστέρηση, 25 λεπτών, γι' αυτό δεν μπορώ να επιτρέψω ε, μπλε κάρτα σήμερα εκτάκτως. Ε. Παρακαλώ, για ένα λεπτό, κύριε Σουρτασούν. Ευχαριστώ πολύ. Βγαίνουμε πιο. μια οικονομική κρίση που σημαίνει σημαντική υποχώρηση των γυναικείων δικαιωμάτων. Η λιτότητα συνδέεται με την πατριαρχική κοινωνία και την άδικη κοινωνία. Και τώρα βλέπουμε να αναδύονται δυνάμεις της ακροδεξιάς που επηρεάζει πάρα πολύ αυτό ε, και στοιχεία του Λαϊκού Κόμματος. Βλέπουμε σαφή επίθεση στα γυναικεία δικαιώματα σε κάποιες χώρες αμφισβητούνται και οι ίδιοι οι νόμοι της έμφυλης βίας, όπως έκανε τώρα η κυβέρνηση στην Ανδαλουσία ή ο πρόεδρος ε, ε, του Λαϊκού Κόμματος στην Ισπανία που θέλει να γυρίσει στο νόμο του 85 για τις αμβλώσεις. Τέτοιες ανισότητες και τέτοια επίθεση υφίσταται γυναίκες. Χρειάζεται μια ατζέντα για την ισότητα, κύριε Επίτροπε, κυρία Επίτροπε, φιλόδοξη, ε, να βγούμε προς τα μπρος επιθετικά με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την κύρωση με κινητοποίηση κινητοποιήσει στο δρόμο και ελπίζω 8 Μαρτίου να είναι μια επιτυχία στις διαδηλώσεις υπέρ των δικαιωμάτων αυτών. Η κυρία Ματέρα, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Φτάσαμε στους τελευταίους μήνες αυτής της θητείας και είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να κάνουμε έναν απαλογισμό όσον αφορά το έργο της Επιτροπής Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά το άρθρο 8 της συνθήκης τελικά δεν εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη, μόλον ότι έχουν ε, καταβληθεί πολύ σημαντικές προσπάθειες. Οι δείκτες για την ισότητα ανδρών και γυναικών δείχνουν ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αποκλήσεις ε, από το 2005 έως το 2015. Και το δεδομένο αυτό μας θλίβει και ουσιαστικά καταδεικνύει ότι θα πρέπει να γίνουν σημαντικές βελτιώσεις σε όλα τα κράτη-μέλη και κυρίως στον τομέα τη απασχόληση, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ σημαντική οπισθοδρόμηση. Βλέπουμε ότι οι γυναίκες πλήττονται ιδιαίτερα σε σχέση με τους άντρε, βρίσκονται σε πολύ πιο επισφαλή θέση και δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή να έχουν υπογράψει όλες οι χώρες τη συνθήκη της ε, Κωνσταντινούπολης. Πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε με πώς είναι ποτέ δυνατόν το ίδιο το Συμβούλιο, μέσα στα πλαίσια του Συμβουλίου να αρνούνται ορισμένες χώρες να προχωρήσουν στην υπογραφή της συνθήκης αυτής. Πρόεδρος, πρέπει να σας πω ότι έχουμε μια καθυστέρηση 25 λεπτών σε σχέση με το αρχικό πρόγραμμα. Ένα μέλος μόνο, μια πολιτική ομάδα μπορώ να δεχθώ πλέον. Σας το λέω αυτό εκ των προτέρων. Η κυρία Σόντροβα, η κυρία Γουόρντ, ο κύριος Γιούρεκ και η κυρία Φορέντσα μόνο, αυτοί που θα μιλήσουν στο, στην, στο στη δικασία Κατστιάι. Η κυρία Χέντα, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Το ζήτημα των δικαιωμάτων των γυναικών και τη προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών από τα ζητήματα με τα οποία έχω ασχοληθεί στο πλαίσιο τη θητεία αυτού του Κοινοβουλίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό να λειτουργεί πραγματικά εύρυθμα Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα τα κράτη-μέλη στα πλαίσια των συνθήκων προβλέπουν εγγυημένα δικαιώματα για τι γυναίκε ή τουλάχιστον αυτό θα πρέπει να ισχύει θεωρητικά. Το πρόβλημα είναι ότι στην πράξη σε ορισμένα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό δεν ισχύει και αυτό πραγματικά με εξοργίζει. Στη δεκαετία αυτή περίοδο που καλύπτει το ψήφισμα αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει μία οργανωμένη με τοπική επίθεση στα δικαιώματα των γυναικών και σαφώ οπισθοδρομούμε. Υπάρχουν συγκεκριμένα πλέον κράτη-μέλη τα οποία περιορίζουν την πρόσβαση στην απορική υγεία προβλέπονται πολλοί περιορισμοί όσον αφορά την απασχόληση των γυναικών και έχουν γίνει ελάχιστες βελτιώσεις μεταξύ του 2005 και του 2015 στον τομέα της απασχόλησης. Για μένα ως φεμινίστρια το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριο Σόλη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. 16,5% η διαφορά στους μισθούς, 40% στις συντάξεις. Μία στις τρεις γυναίκες έχει ε, ζήσει σωματική βία ή σεξουαλική ή και τα δύο. Είναι επίση λιγότερε οι γυναίκες ε, εδώ σε ποσοστό και τα λοιπά. Πάει λέγοντα ο κατάλογος. Ε, πόρο απέχουμε από την πραγματική ισότητα ανδρών και γυναικών. Και ακόμα και αν είναι έτσι, τολμάει η δεξιά κάθε φορά να αμφισβητεί αυτά τα θέματα και κάθε φορά πιο ξαδιάντροπα και πιο ανερυθρίαστα. Ε, πού είναι η προστασία των γυναικείων δικαιωμάτων. Ε, αυτή η δεξιά υπερσυντηρητική νεοφρακική ε, είναι γεγονός στην Ισπανία και αμφισβητεί και την έννοια, την ύπαρξη της φαλοκρατικής ε, ανδρικής βίας. Μιλάνε για ενδοοικογενειακή βία και λένε ότι είναι και ψευδείς οι καταγγελίες. Πού είναι αυτές οι επιθέσεις κατά των δικαιωμάτων απέναντι στις φεμινίστριες. Το έδειξε η 8η Μαρτίου του 18, θα το ξαναδείξει το 19. Η κυρία Σουίτσα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ισότητα ανδρών και γυναικών και τα δικαιώματα των γυναικών ε, είναι από τα βασικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γεγονός ότι διαπιστώνουμε επιστοδρόμηση η υποχώρηση σε ορισμένα γυναικεία δικαιώματα. Εμφανίζονται κάποιες ακραίες τάσεις ε, σε διάφορους κλάδους της κοινωνίας μας. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Η ε, ε, δημοκρατική κοινωνία ε, αναπτύσσεται μόνο εφόσον είναι καλά ανεπτυγμένα και τα γυναικεία δικαιώματα. Συμφωνώ με όσα ακούσαμε και με αυτά που λέει η προφορική ερώτηση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε σήμερα οι γυναίκες να έχουν λιγότερα δικαιώματα από τις μητέρες τους. Τι σημαίνει αυτό. θα πρέπει να πάψουν οι διακρίσεις, οι περιορισμοί των δικαιωμάτων και να ακυρωθεί η σύμβαση ε, της Κωνσταντινούπολης. Υπάρχουν χώρες που έχουν ε, προσχωρήσει σε αυτή τη σύμβαση, αλλά παραμένουν οι ανισότητες και οι διώξεις των γυναικών. Η κυρία Πέτερ, ευχαριστώ πρόεδρε είναι γεγονό πραγματικά ότι η ισότητα ανδρών και γυναικών σήμερα παραμένει ζητούμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να έχουν γίνει κάποιες πρόοδοι στα δικαιώματα των γυναικών, αλλά δεν έχουν διεισδύσει σε όλους τους πολιτικούς θεσμού και παντού στην κοινωνία. Αυτό ισχύει και για την κοινωνική προστασία και σε ό,τι αφορά τη βία κατά των γυναικών. Διακρίσει γίνονται σε διάφορα επίπεδα. Καμιά φορά και πολύ συχνά μάλιστα η γυναίκα θα πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στη σταδιοδρομία, το επάγγελμά τη και την οικογένειά τη. Αντί να μπορεί να τα συμφιλιώνει και τα δύο αυτά. Ε, είναι πολύ σημαντικά τα προβλήματα και δεν σημαίνει ότι οι ορισμοί αλλάζουν και εξελίσσονται ή διαφοροποιούνται ανάλογα με τις μόδες και τους καιρούς και την ιδεολογία. Το αντίθετο, είναι αιώνια αυτά τα δικαιώματα και αρχές. Εγώ αγωνίζομαι ε, για το σεβασμό των δικαιωμάτων κάθε ανθρωπίνου όντως. Και πραγματικά απογοητεύομαι από αυτά που λέει η προφορική ερώτηση και δεν μπορώ να την υποστηρίξω. Σας είπα, για λόγους χρονικούς θα δώσουμε το λόγο σε έναν ομιλητή από κάθε πολιτική ομάδα. Κυρία Σόεντροβα. Ευχαριστώ. Πράγματι, είναι μακρόπνο στόχο η ισότητα μεταξύ των φύλων. Οι διακρίσει ε, είναι ε, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Γι' αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να στηρίξουμε όλα τα μέτρα που θα μας επιτρέψουν να προσεγγίσουμε αυτόν τον στόχο τα δικαιώματα δηλαδή, των γυναικών ε, ε, και το δικαίωμά τους ε, να συμφιλιώνουν τον επαγγελματικό και τον προσωπικό βίο. Οι προτάσεις της Επιτροπής βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, γι' αυτό και τις χαιρετίζουμε. Δυστυχώ ε, βλέπουμε ότι υπάρχει και αρνητική κριτική. Ως μέλος του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματο. μπορώ να πω ότι προστατεύει αυτή η νομική πράξη ε, και τις γυναίκες ε, και τα έμβρια. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε υπέρ τέτοιων πολιτικών. It's είναι σημαντικό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να αντιμετωπίσει αυτή την αρνητική ε, στάση και εναντίωση προ τα δικαιώματα των γενικών, ιδίω εφόσον έχουμε και εκπροσώπου ε, αυτών των απόψεων και εδώ στο Κοινοβούλιο. Βλέπουμε ότι οι στηρητικέ δυνάμει οργανώνονται όλο και περισσότερο, έχουν ε, καταφέρει να πείσουν. όλα ένα και περισσότερο κόσμο λοιπόν ότι αυτοί έχουν δίκιο υπονομεύεται η πρόσβαση ε, των γυναικών ακόμα και στα αντισυλλεπτικά σε κάποιες χώρες. Υπάρχουν εκστρατείε ε, που ε, κινούνται κατά των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ. Είναι πολύ αργή η διαδικασία κύρωση τη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη, παρότι είναι το καλύτερο όπλο για την καταπολέμηση τη ενδοκινιακή βία, η οποία είναι ιδιαίτερα διευρυμένη και εκτεταμένη. Εγώ ανησυχώ για τις εξελίξεις. Ε, υπάρχουν δυνάμει που θεωρούν ότι ο φεμινισμός είναι κάτι το οποίο ανήκει στο παρελθόν. Εμείς όμως πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια και να ε, διαπαιδαγωγήσουμε και τη νέα γενιά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Οι αρχές της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτές οι οποίες πολύ συχνά παραπληροφορούν ε, την κοινή γνώμη. Το άρθρο 14 της Σύμβασης Κωνσταντινούπολης ε, λέει ότι ε, τα σχολεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να προωθήσουν μη τυπικούς και συνθισμένους σεξουαλικούς ρόλους. Ενώ θα πρέπει να προβλέπετε ότι οι γονείς θα μπορούσαν να αντιωθούν σε τέτοιες διδασκαλίες. Επίσης προβλέπονται άλλα σημεία στη σύμβαση αυτή οι, οποία, οι οποίες ουσιαστικά προωθούν διαφορετικές, διαφορετικές συμπεριφορές. Ενδεχομένως να πρέπει να καταργήσουμε ακόμα και την δασκαλία της Οδύσσιας, καθότι εκεί πέρα εμφανίζεται η Πινελόπη να περιμένει για χρόνια ολόκληρα τον Οδυσσέα. Νομίζω ότι στις δικές σας τις χώρες, στη Γερμανία ακόμα έχουμε καταναγκαστικούς γάμους, επομένω σταματήστε να επικρίνετε χώρες όπως η Βουλγαρία, που έχουν πει ότι δεν θέλουν ουσιαστικά τη σύμβαση αυτή. Η κυρία Φορένσα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πραγματικά ότι ζούμε εδώ πέρα μια πολύ σημαντική αντίφαση στην Ήπειρό μας. Από τη μια πλευρά έχουμε ένα κίνημα φεμινιστικό που στρέφεται κατά της σεξιστικής βίας και της πατριαρχικής κοινωνίας και από την άλλη έχουμε συντηρητικά κινήματα. Αναφέρομαι και στη δική μου τη χώρα, δεν ξέρω αν γνωρίζει η Επίτροπος, ότι το Σεπτέμβριο είχαμε την ε, δυνατότητα να ακούσουμε κάποιες ε, Ιταλικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, οι οποίες υπερασπίζουν τα δικαιώματα των γυναικών και οι οποίες δέχονται επιθέσεις από τοπικές Ιταλικές αρχές μη κυβερνητικέ οργανώσει, των οποίων η δράση δεν αναγνωρίζεται και ε, ευτυχώ που τουλάχιστον από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπω άλλωστε έχει πει και η ίδια η Επιτροπή ΦΕΜ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από μια επίσκεψη που έκανε στην Ιταλία, είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προασπίσουμε όλο και περισσότερο το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Ένα δικαίωμα το οποίο ανήκουστο, αλλά αυτή τη στιγμή ακόμα και στην Ιταλία απειλείται. Στην απεργία που θα γίνει στι 8 Μαου θα πρέπει να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο τα δικαιώματα των γυναικών. Η Επίτροπο τώρα έχει το λόγο για να απαντήσει. Αξιότιμα μέλη, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι σας ευχαριστώ για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να προχωρήσει η ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών. Θέλω να αντιδράσω σύντομα, γιατί ξέρω ότι έχουμε καθυστέρηση, ε, να απαντήσω σε δύο μιλητές.